αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος ε, των ορισμών θα ε, επισυναυθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως. Εάν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξουν ενστάσεις, αυτοί οι διορισμοί θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένοι. Τώρα περνάμε στη μέσα διάταξη. Πρώτο σημείο αφορά τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή αναφορικά με την κατάσταση στο κέρα τη Αφρική. Το λόγο έχει έξω του Συμβουλίου ο Υπουργός Αλεξάνδρ Βάνδρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι.